οι αρμόδιες γαλλικές αρχές μας απέστειλαν έτοιμα άρσης βουλευτικής ασυλίας της κυρίας Μιλέν Τροσίνσκι στο πλαίσιο μιας δικαστικής έρευνας, όπως και έτοιμα άρσης ασυλίας του κυρίου Ζαν Μαρί Λεπέν. Στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται, διαβάστηκαν αυτά στην Επιτροπή Νομικών